Τη διάταξη. δήλωση του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ιράν. Δίνουμε το λόγο λοιπόν στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, στον κύριο Καρλ Μπίλτ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή γιατί για πρώτη φορά έρχομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρώτη, αλλά όχι και τελευταία. Θα έρθω πολλές φορές στο επόμενο εξάμεινο για να συζητήσουμε πολλά θέματα. Και αυτή τη φορά το θέμα που μας αφορά είναι το Ιράν. Πριν επισέλθω στην ουσία του θέματος, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για το τραγικό δυστύχημα που ενέσκυψε σήμερα. Λυπούμαστε ειλικρινά για όσους έχασαν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους. Το θέμα του Ιράν είναι πολύ σημαντικό στην, στο πρόγραμμα εργασιών της, Ευρω... της Σουηδικής Προεδρίας. Έχει σχέση με τις εκλογές και τα ερωτηματικά καταφημισμών, ας πούμε, που προέκυψαν μετά τις εκλογές, καθώς και τις πολιτικές εξελίξεις που έλαβα χώρα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ευρωπαϊκή θέση ήταν πολύ αποφασιστική και κατηγορηματική για τις εκλογές στο Ιράν. Είπαμε ότι διαφιλονικές ε, περί της έκβασης των εκλογών ε, θα πρέπει να διερευνηθούν από τις Ιρανικές αρχές. Βέβαια, γίναμε μάρτυρες των ε, γεγονότων στους δρόμους της Τεχεράνης και καταδικάσαμε τη χρήση βίας, την επίδειξη ισχύω έναντι ειρηνικών διαδηλωτών, τις καταδίκες δημοσιογράφων, τις απελάσεις δημοσιογράφων, τις καταπιέσεις των διαδηλωτών. Αυτές οι συμπεριφορές όχι μόνο αντιβαίνουν στις δικές μας αρχές και αξίες, αλλά δυστυχώς διαψεύδουν τις προσδοκίες μας για μια πιο ανοιχτή, διαφανή και δημοκρατική κοινωνία στο Ιράν, στην οποία προσβλέπουν πολλοί Ιρανοί πολίτες. Το Ιράν εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής μας. Θέλουμε νέες και καλύτερες σχέσεις με το έθνος του Ιράν, γιατί πιστεύουμε ότι το έθνος του Ιράν μπορεί να συμβάλλει στις γενικότερες εξελίξεις παγκοσμίω, αλλά και στις εξελίξεις στην περιοχή. Και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει δυνατότητα για μια ανανέωση των σχέσεών μας με το Ιράν. Και πριν ολοκληρώσω θα ήθελα να επισημάνω ένα θέμα που μας απασχόλησε αρκετά. Οι Ιρανικές αρχές προέβησαν σε κρατήσεις πολλών ε, προσωπικότητων που ήταν υπάλληλοι ευρωπαϊκών αποστολών και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι επίκοοι. Έχουμε συνεχείς επαφές με τις Ιρανικές αρχές και πραγματοποιούμε διαβήματα για το θέμα αυτό και οι κατηγορίες ε, που απαγγέλθηκαν κατά των ε, Ευρωπαίων αυτών είναι ανεδαφικές, ανυπόστατες. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαθετήσουμε αυτό το θέμα με τις Ιρανικές αρχές και να φέρουμε σε αίσιο πέρα στην αποστολή μας, δηλαδή να οδηγήσουμε στην απελευθέρωση αυτών των υπαλλήλων. Ευχαριστώ κύριε Μπίλτ. Η Επίτροπος, η κυρία Άστον, έχει το λόγο για ένα πεντάλεπτο. Προφανώς θα επιδείξουμε και κάποια ευελιξία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτη με ευκαιρία να συγχαρώ όλα τα αξιότιμα μέλη για την εκλογή τους στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκ μέσω Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να πω ότι Προσβλέπουμε σε επικοδομητική συνεργασία μαζί σας και θα αντιμετωπίσουμε μερικές πιεστικές ε, προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Το θέμα της συζήτησής μας σήμερα είναι ένα από τα προβλήματα αυτά. Η κυρία Μπενίτο Φεραίρο Βάλτον, η συνάδελφός μου, ταξιδεύει αυτή την εβδομάδα και προσφέρθηκα με χαρά να μπορέσω να μιλήσω εκ μέρους της στο Κοινοβούλιο σήμερα. Αυτό το Κοινοβούλιο διαδραματεί σημαντικό ρόλο διατηρώντας και αναπτύσσοντας σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Γίνονται επισκέψεις της αντιπροσωπείας ε, του Κοινοβουλίου για το Ιράν και έρχονται και εκπρόσωποι του Ιράν εδώ και οπότε έτσι αναπτύσσεται αμοιβαία κατανόηση. Το Κοινοβούλιο έπαιξε το ρόλο του δημιουργώντα ε, δημιουργώντας διάφορα μέσα που είναι σημαντική βάση για δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ιράν και εμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζουμε να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε καλά αυτά τα μέσα στα επόμενα χρόνια. Η σημερινή συζήτηση ξεκίνησε από τις πρόσφατες Ιρανικές προεδρικές εκλογές και τα γεγονότα που ακολούθησαν. Όπως είπε η Προεδρία, οι εξελίξεις των πολιτικών στο Ιράν είναι θέμα βασικά που αφορά τους πολίτες του Ιράν. Αλλά έχουν ευρύτερη σημασία αυτά τα γεγονότα και πρέπει να ακολουθούμε εκ του σύνεγγυ τη εξελίξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τοποθετήθηκε σαφέστατα όσον αφορά την κατάσταση στο Ιράν μετά τι προεδρικέ εκλογέ και παρέμεινε ενωμένη στη θέση της αυτή. Εκφράσαμε πλήρη σεβασμό όσον αφορά την κυριαρχία του Ιράν, αλλά τονίσαμε τη μεγάλη μας ανησυχία, βαθιά ανησυχία για τα βία επεισόδια που ακολούθησαν τις εκλογές, όπω θα κάναμε πάντα όταν διακυβεύονται δικαιώματα ή χάνονται ζωή σε οποιαδήποτε χώρα. Οι εικασίε ευρωπαϊκή παρέμβαση σε εκλογέ στο Ιράν ή ασδήποτε ανάμειξη στι διαμαρτυρίε που ακολούθησαν είναι κάτι αβάσιμο. Όμω, η καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων ε, δημιουργούν εντάσει. Και η φήμωση των μέσων είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αυτά δεν είναι θέματα που περιορίζονται στα εσωτερικά ή ασδήποτε χώρας. Παρά την ευαισθησία της καταστάσεω στο Ιράν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει πραγματικά ότι θα πρέπει να παραμείνει να διατηρηθεί ο διάλογος. Αυτό ίσχυε και πριν τις εκλογές και εξακολουθεί να ισχύει και τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράν έχουν πολλά κοινά σημαντικά συμφέροντα, όπως είναι η καταπολέμηση τη διακίνηση ναρκωτικών και η υποστήριξη των προσφύγων των Αφγανών. Αυτά είναι θέματα που χρειάζονται συνεχή προσοχή και συνεργασία και ελπίζουμε να συμμερίζεται αυτή την άποψη του Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να προσπαθεί να βρει τρόπο για τη χρήση κοινοτικών μέσων σε επικοδομητικές δραστηριότητε στο Ιράν. Μπορούμε να αυξήσουμε την αμοιβαία κατανόηση συνεχίζοντας τη συνεργασία μας, παραδείγματος χάρη μέσω του Erasmus Mundus, των πανεπιστημιακών ανταλλαγών. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κρατήσει όλες τις, διά, όλους τις διάβλους ε, επικοινωνίας με το Ιράν ανοιχτέ. Θα πρέπει ε, να συνομιλούμε το Ιράν σε όλα τα επίπεδα όποτε είναι δυνατόν και θα πρέπει να συνεχίσουμε όποτε αυτό ε, αρμόζει τη συνεργασία στο μέλλον. Οι παρούσες διαφορές μας στην κυβέρνηση του Ιράν είναι πολλές. Κάποιες από αυτές τις διαφορές είναι σοβαρότατες. Καλούμε την κυβέρνηση του Ιράν να έρθει κοντά μας, να προσπαθούμε να βρούμε ε, λύσεις στις διαφορές μας μέσω διαλόγου. Μόνο μέχρι συζητήσεων των προβλημάτων που έχουμε μεταξύ μας, με αμοιβαίο σεβασμό μπορούμε να ελπίσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Η Ευρώπη ποτέ δεν έκλεισε την πόρτα σε τέτοιες συζητήσεις και εξακολουθεί να είναι ανοιχτή και σήμερα. Και τέλος, Πρόεδρε, όπως και η Προεδρία, θέλω να εκφράσω τη συλληπιτήριά μου για τις οικογένειες των Ιρανών και των Αρμενίων θύματα του τραγικού γεγονότος του αεροπορικού δυστυχήματος που συνέβη σήμερα. Grazie. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε. Και τώρα ξεκινάει η συζήτηση. Ο κύριος Σάρος Βόλσκι έχει το λόγο για δύο λεπτά. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σα αναφέρω ότι έγινε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων την τελευταία Τετάρτη γιατί η νέα σύσταση της Επιτροπής δεν έχει ακόμα συνέλθει. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τα γεγονάτα. Δεν θα πρόκειται λοιπόν να αναφερθώ σε αυτό. Η Ένωση θα πρέπει να τονίσει την καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να παρακολουθήσει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον Ιράν και να καλέσει το Ιράν ε, να απολογηθεί για τη βία που παρουσιάζεται. Εμείς ε, συναντηθήκαμε με τους αντιπροσώπους της ε, κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν και νομίζω ότι αυτή η πτυχή είναι εξαιρετικά σημαντική. Συμφωνούμε τις ε, τοποθετήσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Καλούμε όμως το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι τηρούνται στην Τεχεράνη οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι δεν λαμβάνουν χώρα βασανιστήρια. Θα πρέπει επίσης να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επιμένουμε να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέτρα για να υποστηριχθεί η κοινωνία των πολιτών στην στο Ιράν. Όχι μόνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την δημοκρατία, για το κράτος δικαίου για να καταπολεμηθούν το λαθροπόριο ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων, για να αναφέρουμε μερικά από τα εγκλήματα. Γιατί αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει την ελευθερία του λόγου στη χώρα. Να ασκήσουμε πίεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ναι, αλλά όχι με τίμημα την απομόνωση, γιατί θα πρέπει να υπάρξει διάλογος ακόμα και αν είναι δύσκολος. Διανύουμε μια πολύ δύσκολη, ε, δύσκολη περίοδο στο Ιράν για θέματα πρινικά, για παράδειγμα των Και αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η συνέχεια. Πιστεύουμε ότι η Ένωση θα πρέπει να βρει έναν τρόπο για να ξαναξεκινήσει το διάλογο με το Ιράν για τα πολύ σημαντικά αυτά θέματα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέα εμπιστοσύνη και να ξεκινήσει μια νέα οδός διπλωματικής επικοινωνίας και επίσης θα υποστηρίξουμε το Συμβούλιο και την Επιτροπή στην προσπάθεια αυτή και εσωτερικά στο Κοινοβούλιο θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να βελτιωθούν οι διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν. Ευχαριστώ κύριε Σάιρο Βούλσκι που μίλησε εν ονόματι της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δίνουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ο κύριος Χόβιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ό,τι και να αισθάνονται οι άνθρωποι για τα αποτελέσματα των ελληνικών εκλογών, δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι δεκάδες και εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, δεκάδες σκοτώθηκαν στις διαμαρτυρίες που έγιναν μετά τις εκλογές στη χώρα και χιλιάδες άνθρωποι κρατούνται ως πολιτικοί κρατούμενοι. Και όλο το Κοινοβούλιο χωρί δισταγμό θα πρέπει να καταδικάσει αυτές τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα πρέπει να καταδικάσει και την παρεμπόδιση τη ελευθεροτυπίας που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των εκλογών. Όπω είπε και ο Σαροσβόλσκι, από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων την περασμένη εβδομάδα και εμεί να αναγνωρίσουμε ότι καλύτερος τρόπος, ένας από τους καλύτερους τρόπους για να καθοριστούν οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές είναι να κληθούν παρατηρητέ να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολύ καλό ιστορικό σε αυτό το θέμα και θα πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρου μα δεν πίστευε ότι θα μπορέσει να κάνει αντικειμενική και δίκαιη δουλειά όσον αφορά τι εκλογέ. Και μπορούμε να πούμε γι' αυτό ότι δεν έχουμε και εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα των εκλογών. Πρόεδρε, η καρδιά μα στρέφονται προς τους Ιρανούς που κρατούνται και που παραδιάστηκαν τα δικαιώματά τους. Οι σκέψεις μας είναι μαζί τους πάνω απ' όλα. Ζητώ από το Κοινοβούλιο να στείλει τις σκέψεις μας και τον Ιρανό υπάλληλο της Βρετανικής Πρεσβείας που κρατείται και κατηγορείται ότι παρακινούσε τις διαδηλώσεις με αβάσιμο τρόπο και θα πρέπει να φτάσουμε την υποστήριξή μας και στο Γάλλο φοιτητή που φυλακίστηκε από τις Ιρανικές αρχές και θα πρέπει να επενέσουμε τους συναδέλφους Σουηδικής Προεδρίας που υποστήριξαν αυτούς τους ε, ανθρώπους ε, και συντονισμένα κινήθηκαν από την τη Ευρωπαϊκή Ενώση, θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Λυπούμε που το Ευρωπαϊκό Εθνικό Κύμα μίλησε για πρώτη φορά και ο βουλευτής είπε ότι το Ισλάμ είναι ένα, ένα καρκίνωμα που θα πρέπει να αφαιρεθεί μέσω χημοθεραπείας από την Ευρώπη. Αυτό δεν εκπροσωπεί τους Βρετανούς, δεν είναι η στάση της Ευρώπης όσον αφορά το Ισλάμ και θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή τη θέση όπως ε, αντιστεκόμαστε και σε διάφορες ειδικέ που συμβαίνουν διεθνώς. Ευχαριστώ κύριε Χάουιτ και τώρα να δώσουμε το λόγο για τη συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη Σνέιτς Ούτεμπεκ είναι το επόμενο όνομα. Η κυρία Νέιτς. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Ιράν αποτελεί, είναι μια μεγάλη χώρα με μεγάλο και κυρίως νεαρό πληθυσμό και μεγάλη ιστορία και πραγματικά εντυπωσιακό πολιτισμό. Το Ιράν επιπλέον αποτελεί και μια χώρα σε μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές του κόσμου. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει και για λόγους ανθρωπιάς να, να μην μας αφήνει αδιάφορους η κατάσταση στο Ιράν. Δεν είμαστε υπέρ της ε, αναγκαστικής αλλαγής καθεστώτος. Ωστόσο, θεωρούμε ότι όλοι οι λαοί του κόσμου και ο λαός του Ιράν θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν τους πολιτικούς τους ηγέτες και να τους αλλάζουν όποτε θεωρούν ότι δεν, ε, επαρκούν τις, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις οι εκλογές στο Ιράν δεν πληρούν τους όρους για τις δίκαιες εκλογές, τα παγκόσμια, τέτοια, τα παγκόσμια αυτά ε, πρότυπα. Και αυτό συνέβη και στις τελευταίες εκλογές, αλλά μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στο Ιράν δεν αποδέχθηκαν το εκλογικό αποτέλεσμα και βγήκαν στους δρόμους. Οι πολλοί υπομονετική αναθεώρηση του εκλογικού αποτελέσματος δεν έπεισε τα πλήθη αυτά και γι' αυτό λοιπόν συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις. Οι διαδηλώσεις αυτές ε, καταστάθηκαν με πολύ βιαίο τρόπο και συνεχίζονται οι διώξεις. Και εμείς κατηγορούμε τις ε, διώξεις αυτές, καταδικάζουμε τις διώξεις αυτές και καλούμε τις Ιρανικές αρχές να απελευθερώσουν όλους τους φυλακισμένους και να σταματήσουν τις ε, διώξεις και η δίωξη των ε, αλλαταπών δημοσιογράφων και του διπλωματικού προσωπικού θα πρέπει να σταματήσουν επίσης άμεσα. Συνάδελφε, πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα, πρόεδρε της Επιτροπής, τα καθεστώτα που ανατρέπονται με τον τρόπο αυτό και στρέφονται κατά του ίδιου του πληθυσμού τους, κατά της, των ίδιων τους των νέων, χάνουν πάσα νομιμότητα, όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Και είναι ιδιαίτερα τραγικό ότι το δράμα αυτό λαμβάνει η χώρα μια στιγμή που ο πρόεδρος των ε, Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να ξεκινήσει διάλογο. Το Ιράν ε, πρόκειται να χάσει μια ιστορική ευκαιρία σε παγκόσμιο προσκήνιο, να χάσει τη θέση που αναλογεί στην ιστορία της και στον πολιτισμό τους. Σας ευχαριστώ κυρία μου και γιατί τηρήσατε το χρόνο που ήταν στη διάθεσή σας. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Κον Μπέντιτ που είναι πρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων και θα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε, Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε εύοντα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν ένα έθνος θέλει να απελευθερωθεί πραγματικά είναι άξιο θαυμασμού και άξιο της αλληλεγγύης μας. Και αυτό ισχύει τώρα με τον Ιρανικό λαό. Ούτως ή άλλως ήταν ε, νοθευμένες οι εκλογές από τη βάση τους. Αλλά ακόμη και σε αυτές τις εκλογές είδαμε ότι ο Ιρανικός λαός βρήκε ένα ρήγμα, ένα κενό για να μπορέσει να εκφράσει τη βούλησή του για ελευθερία και δημοκρατία. Φυσικά έχουμε συμφέροντα, φυσικά θέλουμε να συνεχιστεί ο διάλογος με το, με την τρομοκρατική ιρανική εξουσία, αυτό δεν το αφισβητεί κανεί, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να, συ, συζητούμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτά που συνέβησαν στην Τεχεράνη είναι αποτρόπαια. Καθημερινά γίνονται βασανιστήρια στις Ιρανικές φυλακές. Δεν βασανίζονται μόνο Βρετανοί υπήκοοι, αλλά και Ιρανοί υπήκοοι και οι γυναίκες από το Ιράν καθημερινά υφίστανται βασανιστήρια στις Ιρανικές φυλακές. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να υψώσει τη φωνή της. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των ε, συμφερόντων του Ιρανικού λαού και τη πρόάσπιση των συμφερόντων του και των δικών μας συμφερόντων που δεν συμπίπτουν πάντα με αυτά του Ιρανικού λαού. Η κατάσταση είναι περίπλοκη, αλλά θα πρέπει να διατρανώσουμε την υποστήριξή μας προς τον Ιρανικό λαό. Θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσω το θέμα της συμμετοχής και της, της και της Siemens στην καταστολή του Ιρανικού λαού και την ευθύνη που έχουν ε, ευρωπαϊκές βιομηχανίες οπλισμού ε, για την καταστολή αυτή. Γιατί οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, επέτρεψαν στην Ιρανική κυβέρνηση να καταπιέσει τον Ιρανικό λαό και να καταστήλει την ελευθερία του. Ευχαριστώ κύριε Κονμπεντίτ. Οικονομήσατε και 10 δευτερόλεπτα, μίσατε λιγότερο. Ο κύριος Στίβενσον έχει το λόγο. Τη ομάδα των συντηρητικών μεταρρυθμιστών, Ευρωπαίων μεταρρυθμιστών. Έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, ενώ καθόμαστε εδώ και συζητάμε την εξέγερση την πρόσφατη στο Ιράν, καταλαβαίνουμε ότι πάνω από 50 ηγέτες των σπουδαστών κρεμάστηκαν από τις αρχές. Πάνω από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στους δρόμους και ΝΕΝΤΑ που έγινε διεθνές σύμβουλο, σύμβολο. Η ΝΕΝΤΑ που έγινε σύμβολο, σύμβολο της καταπίεσης του φασιστικού αυτού καθεστώτος. Και ενώ εξακολουθούμε να απολαμβάνουμε τη θέση που έχουμε σαν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος με την Ιρανική κυβέρνηση θεωρούμε σοβαρά ότι τα χρήματα είναι σημαντικότερα από τις ζωές γιατί δεν επιβάλλουμε ε, πιο σοβαρές κυρώσεις. Εμείς, σαν κοινοβούλιο, γιατί δεν καταργούμε την αντιπροσωπεία μας για σχέση με το Ιράν, που ούτως ή άλλως την τελευταία πενταετία δεν έγινε τίποτα άλλο παρά ένα αφαιρέφωνο της Ιρανικής πρεσβείας στην, ε, στις Βρυξέλλες και ντροπιάζει τα ευρωπαϊκά θεσμικά οργάνα. Την καταργήσουμε, να μιλήσουμε σκληρά στις Ιρανικές αρχές. Αυτή είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Ευχαριστώ κύριε Στέβενσον. Δίνουμε το λόγο τώρα στον κύριο Σόλτς της Ενωτικής Αριστεράς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η γκουε NGL ανησυχεί ιδιαίτερα για την συνεχιζόμενη βία που παρουσιάζεται στο Ιράν και εμείς καταδικάζουμε τις ε, παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των διαδηλωτών. Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση των ε, κρατουμένων και θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να το απαιτήσει αυτό από κοινού. Επίσης, ε, επικρίνουμε τα σχόλια ε, του τύπου και των κυβερνήσεων που χρησιμοποιούν το νόμιμο δικαίωμα των διαδηλωτών. Η ομάδα μου καταδικάσει τις στρατηγικές αυτές και γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζουμε τα σαφή λόγια του Ομπάμα για να μην δοθεί στο Ισραήλ πράσινο φως για την εισβολή στο Ιράν. Και ο Αμερικάνος ε, πρόεδρος χρησιμοποιεί τη διπλωματία. Είναι κυρίαρχο κράτος το Ιράν και μόνο ο ίδιος ο λαός του Ιράν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση ενός κυρίαρχου κράτους θα πρέπει να ακολουθεί τις επιθυμίες του λαού. Σας ευχαριστώ κύριε Σόλτς. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον επόμενο στον κατάλογο προβέρα της Ευρώπης των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας που έχει 1,5 λεπτό ο κύριος Προβέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Η καταστολή των πολιτών που διαμαρτύρονται και αμφισβητούν τα αποτελέσματα των εκλογών, η λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης η δίωξη της αντιπολίτευσης επιβεβαιώνουν την έλλειψη δημοκρατίας στο Ιράν. Αν όλες καταστάσεις ε, υπάρχουν και σε άλλες χώρες όπως είναι η Κίνα, αλλά για το Ιράν υπάρχουν και άλλοι λόγοι για να ανησυχούμε. Πρώτος λόγος, οι γεμονικές φιλοδοξίες που εκδηλώνονται μέσω της αναμίξεως σε γειτονικέ χώρες. Στην περιοχή της Βασόρα στο Ιράκ, η υποστήριξη της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Δεύτερος λόγος, η μεγάλη επιρροή του θρησκευτικού εξτρεμισμού που ασκεί στην πολιτική εξουσία, στην Ισλαμική Δημοκρατία. Πριν από λίγε ώρες ένα τραγουδιστή καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια ε, διότι πρόσβαλε την θρησκεία και 12 Σουνίτες καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο πρόεδρος Αχμαντινετζάντ επανειλημμένα διακήρυξε ότι η καταστροφή του κράτους του Ισραήλ είναι στόχος προτεραιότητας για την πολιτική του. Και η βούληση του Ιράν να αναπτύξει ένα πυρηνικό πρόγραμμα είναι ανησυχητικό πράγμα. Και μάλιστα εκτό των διεθνών ελέγχων. Θεωρώντας ότι η Ιράν είναι ένα από του μεγαλύτερου παραγωγού φυσικού και πετρελαίου, πραγματικό στόχο, είναι η ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων για να μπορεί να εκβιάζει τι χώρε τη περιοχή και όλη την διεθνή κοινότητα το Ιράν. Χρειάζεται λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια από πλευρά ευρωπαϊκή πολιτική για να βρεθεί σωστή ισορροπία. Δηλαδή, έχουμε από τη μια πλευρά την, ηγεσία των Χεσμολά και από την άλλη έχουμε την μεταρρυθμιστική πτέρυγα του Ιράν που υπάρχει. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των δύο πλευρών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οικονομικού πόρου για αυτόν τον σκοπό το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για να υποστηρίξουμε όλα τα θύματα τη καταστολή και τη καταπίεση. Καμία πολιτική παρέμβαση μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρί να είναι ενωμένη και κοινή η δράση και να συμφωνούν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Προβέρα. Και το λέω όχι μόνο για αυτά που είπατε, το ευχαριστώ. Μάλλον ότι αν ξεπερνάτε, δεν το λέω μόνο για σας, δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα όρια. Δεν μπορούμε να ξεφεύγουμε πάνω από μισό λεπτό όταν σας δίνουμε ένα μισή λεπτό. Σας το λέω με κάθε ευγένεια, κύριε Προβέρα. Δεν αναφέρομαι σας προσωπικά που ξεπεράσετε το χρόνο σας, αλλά γενικά μιλάω. Η κυρία Χριστίνα Μορβάη έχει το λόγο, των μη εγγεγραμμένων, ε, για δύο λεπτά. Thank Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως ε, δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με 20 ετή πείρα διεθνώς στον τομέα αυτό, θα ήθελα να θέσω μια έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να έχουμε νομιμοποίηση και αξιοπιστία για τον έλεγχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τρίτο κόσμο και σε εξωκοινωτικέ χώρες, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε τα του οίκου μας και να δούμε πώς έχει η κατάσταση τη δημοκρατία, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στη δική μου την πατρίδα, την Ουγγαρία. Θα σας δώσω ορισμένα στοιχεία. Στις 23 Οκτωβρίου του 2006 οργανώθηκε μια σημαντική διαδήλωση με 100.000 περίπου άτομα για την επέτειο της ε, επανάστασης ε, του 1956 οργανώθηκε από το ΦΙΝΤΕΣ, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, που εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα κέρδισε τις ε, εκλογές φέτος στην Ουγγαρία. Ήταν ε, ένα πλήθος ε, μεσοστικών οικογενειών με παιδιά και μάλιστα η η ουγγρική αστυνομία επιτέθηκε σε αυτό το πλήθος με δακρυγόνα προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς εκατοντάδων ανθρώπων. Και την ίδια ημέρα εκατοντάδες άνθρωποι φυλακίστηκαν παράνομα και βασανίστηκαν στις ουγγρικές φυλακές. Έκτοτε και τα τελευταία τρία χρόνια, μέχρι πρόσφατα, όπου είχαμε 216 ειρηνικούς διαδηλωτές ε, συνελήφθησαν και αυτοί παράνομα και κακοποιήθηκαν από την αστυνομία. Πολύ συχνά μέσα σε αυτή την τριετία όταν διοργανώνονταν αντικυβερνητική διαδήλωση, δεν μιλούμε για το Ιράν, την Κίνα και την Ονδούρα, μιλούμε για μια κοινοτική χώρα, την Ουγγαρία. Τα ίδια πράγματα συμβαίνουν. Μαζική χρήση βία, κακοποίηση και βαρβαρότητε, βαναυσότητε από πλευρά αστυνομία μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άσχετα με την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκει ο καθένα. Θα πρέπει να διερευνήσει την κατάσταση αυτή, να βρει του υπετίου, να απονεμηθεί δικαιοσύνη για τα θύματα και να σταματήσει αυτή η μαζική και κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι θα αποκτήσουμε την αξιοπιστία και θα έχουμε την ομοποίηση για να ελέγχουμε την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν ή οπουδήποτε αλλού εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μόρβαη. Το λόγο έχει ο κύριος Μίλαν Μον για δύο λεπτά. Εγώ θα μιλήσω για το Ιράν, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω και εγώ τα συλληπιτήριά μου για το αεροπορικό δυστύχημα που ενέσκυψε σήμερα το πρωί. Εστερνίζομαι πολλές ε, από τις ιδέες που ακούσαμε για το Ιράν μετά τις ε, εκλογές που δεν ήταν ούτε ε, ελεύθερες ούτε ανώθευτες και επέτρεψαν ε, τον αχματινετζάν να παραμείνει στην εξουσία καταπιέζοντας τους διαδηλωτές, ε, τους ε, αντιφρονούντες, τους δημοσιογράφους και μάλιστα η εξουσία αυτή χρησιμοποιεί και την παραπληροφόρηση για να χειραγωγήσει το κοινό. Βέβαια, το καθεστώς του Ιράν έχει υποβαθμιστεί και στο εσωτερικό αλλά και η εικόνα του στο εξωτερικό έχει αμαυρωθεί. Και νομίζω ότι θα τροποποιηθεί και η κατάσταση εντός του καθεστώτος. Ιδιαίτερα αν δεν ανεβούν οι πετρελαϊκές τιμές και δεν βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να συνεχίσει να καταδικάζει τις καταχρήσεις που διαπράττονται στο Ιράν, να ζητήσει μεγαλύτερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών, τον άμαχο πληθυσμό, και κυρίως τους Ιρανούς που είναι υπέρ της δημοκρατίας, του πλουραλισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν θα πρέπει να απογοητεύσουμε αυτά τα στρώματα της κοινωνίας που προσβλέπουν στη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δούμε και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που αποσταθεροποιεί την περιοχή αλλά και αντιβαίνει στο γενικό πρόγραμμα τη μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων. Χαίρομαι που το Ιράν είναι προτεραιότητα τη Σουηδική Προεδρία. Θα πρέπει στη συνεργασία να συμπεριλάβουμε και τη Ρωσία και την Κίνα που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία. Η υποστήριξή του είναι απαραίτητη για να βρούμε μια συνενετική λύση για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη απειλή ε, που απαιτεί μια αποφασιστική στάση από την παγκόσμια κοινότητα. Και συμφωνώ με το ψήφισμα που εθέτησε η G8 την περασμένη εβδομάδα. Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων κατέδειξαν τον εξτρεμισμό, το ριζοσπαστικό χαρακτήρα και τη στάση των Ιρανών ηγετών. Είναι σαφές ότι η παγκόσμια κοινότητα δεν μπορεί να επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλα. Σας ευχαριστώ. Μονή για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσω την παρθενική μου ομιλία στην Ολομέλη αυτή, εκφράζοντας την ικανοποίησή μου που η συζήτηση αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν δεν προκλήθηκε μόνο από την κατάσταση μετά τις εκλογές. Γιατί η πρόσφατη εκτέλεση Σουνιτών στο Ιράν επανέφερε τη χώρα αυτή στην επικαιρότητα και στους πηχαίους τίτλους των, του διεθνούς τύπου. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο το πρόγραμμα της εξωτερικής μας πολιτικής. Μιλούμε για το Ιράν και τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί θέλουμε μια συνεπή και σοβαρή αντιμετώπιση του ρόλου μας ε, στις εξωτερικές υποθέσεις και ιδιαίτερα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάτι τέτοιο, κύριε Πρόεδρε, προϋποθέτει τη συνεπή χρήση όλων των μηχανισμών και εργαλείων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Και στην περίπτωση του Ιράν δεν θα πρέπει να έχουμε στεγανοποίηση των διαφόρων τομέων του διαλόγου. Ο διάλογος για, για τα πυρηνικά δεν θα πρέπει να γίνεται ερήμη του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί ο διαρθρωτικός διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει διακοπεί από το 2004. Δεν υπάρχει συμφωνία συνεργασίας και εμπορίου για να μπορέσουμε να προσθέσουμε εκεί μια δημοκρατική ρήτρα. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια για την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που δυστυχώς είναι πενιχρά. Θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη χρήση των μηχανισμών που έχουμε στη διάθεσή μας. Κάποιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και από την Ιρανική Αντιπολίτευση ζήτησε απόλυτη διακοπή των σχέσεών μας με το Ιράν και μία αναγνώριση της νέας κυβέρνησης. Εμείς καταδικάζουμε απερίφραστα την πολιτική καταστολή και τη φήμωση της ελεύθερης έκφρασης στο Ιράν, αλλά δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχνούμε την προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας στην περιοχή αυτή, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό χρειαζόμαστε διάλογο, διπλωματία, αναζήτηση κοινών συμφερόντων και σφυριλάτηση μια συμμαχία των πολιτισμών. Αυτή την έκκληση θα ήθελα να απευθύνω προς το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία μου. Τώρα, το επόμενο όνομα που έχουμε μπροστά μας είναι Ρόσμπαχ, για ένα λεπτό. Κυρία Ρόσμπαχ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα συζήτησε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Και ξανά αυτό κάνουμε σήμερα. Εξετάζοντας το θέμα, Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι απτό επιτέλους. Μιλάμε για ανθρώπους που διψούν για ελευθερία και βγαίνοντα στους δρόμους προσπάθησαν ε, να ρίξουν ένα εγκληματικό καθεστώς. Είναι ένα καθεστώς που δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα. Θα πρέπει να δούμε τι ρόλο έχει διαδραματίσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πρέπει αυτοί που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα να απολογηθούν. Ο κ. Αχμαντινετζάτ θα πρέπει να δικαστεί από διεθνές δικαστήριο. Θα πρέπει να δούμε πόσο η ΕΕ μπορεί να υποπτεύει τις ελευθερίες. Στην τελευταία συνεδρία της αντιπροσωπεία για το Ιράν μετατράπηκε σε ένα εργαλείο ε, για το Ιρανικό καθεστώς δεν μπορούμε να συνεργαζόμαστε με δικτατορία. Σε ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Να δώσουμε το λόγο στον επόμενο αγορητή, Γκρίφιν, για δύο λεπτά. Κύριος Γκρίφιν. Πρόεδρε, ήμουν παρατηρητής ε, στις ε, διαδηλώσεις του για την ε, Επανάσταση του 1956 στη Βουδαπέστη και έχει δίκιο η συνάδελφο ότι καταδικάζουμε την κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζονται στο Ιράν και αγνοούμε τι ανάλογε καταστάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναρωτιέμαι αν θα είμαστε αρκετά υποκριτικοί για να καταδικάσουμε το Ιράν για τη χρήση βία στι εκλογέ όταν ο Ντέβιτ Κάμερον είναι από του σπόνσορες του UAF, μια οργάνωση ακροδεξιών εγκληματιών που χρησιμοποιεί βία κατά των ε, εθνικών ε, αντιφρανούντων στην Βρετανία. Και οι, οι ίδιοι βουλευτές ε, στην Αγγλία χρησιμοποιούν τη φορολογία του πολίτη στη Βρετανία για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις δράσεις τους. Το βασικό στοιχείο όμως που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξή. Μπορεί να είμαστε καλοπροαίρετες ε, οι κριτικές μας προς το Ιράν και δικαιολογημένε, αλλά θα χρησιμοποιηθούν ως προπαγάνδα πολεμική από τα κατεστημένα για την ε, που έχουν συμφέροντα για την ε, στρατιωτική επέμβαση στη χώρα αυτή οι πετρελαϊκές εταιρείες και όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να καταστραφεί την κυριαρχία του Ιράν από έναν επιθετικό πόλεμο. Ούτε οι φιλελεύθεροι οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να πιστέψουν ξανά το ψέμα των πρινικών όπλων. Άρα χρησιμοποιούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα ως νέα δικαιολογία. Ας μην προσθέσουμε τη φωνή του οίκου μας για μια τρίτη παράνομη και αντιπαραγωγική ε, επίθεση του δυτικού κόσμου προς την ε, προς τον ε, μουσουλμανικό κόσμο. Για να μην χρησιμοποιήσουμε τα 18χρονα βρετανικά αγόρια από τη να, καλέσουμε, να τους καλέσουμε να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους τα παιδιά για να τα στείλουν στον πόλεμο ή αλλιώς να κοιτάξουν τη δουλειά τους. Ευχαριστώ. Κύριε Γκρίφιν, και τώρα επόμενος αγορητής Κασμάρε, κύριος Κασμάρεκ δύο Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ο θάνατος αθώων είναι πάντα τραγικός. Όταν όμως χάνονται στο βωμό της υπεράσπισης σημαντικών αξιών όπως είναι η ελευθερία και η δημοκρατία, τουλάχιστον δεν πάει χαμένος, δεν είναι μάταιος αυτός ο θάνατος. Το Ιράν συλλαμβάνει παράνομα, βασανίζει και σκοτώνει ε, τους διαδηλωτές. Δεν υπάρχει ελευθερία έκφραση. Θα πρέπει λοιπόν η κοινή γνώμη να αντιληφθεί την πραγματική φύση του Ιρανικού καθεστώτο. Ε, είναι ένα καθεστώ που απέχει πόρο από του ουσιαστικού ε, κανόνε και τι ελάχιστε προδιαγραφέ τη παγκόσμια κοινότητα. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση που είναι απαράδεκτη. Βέβαια, σε τέτοιε περιπτώσει ανακύπτει το γνωστό ερώτημα. Τι μπορούμε να κάνουμε μπορούμε να υποστηρίξουμε τις προτάσεις που ήδη διατυπώθηκαν. Καταρχήν, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να σταματήσουν να χρησιμοποιούν βία έναντι όσων διαφωνούν με τις δικές τους απόψεις. Θα πρέπει να να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και η παρακολούθηση του σεβασμού αυτού να εξασφαλιστεί από την παγκόσμια κοινότητα. Επίση, θα πρέπει να διεξαχθούν ελεύθερε και ανώθευτες εκλογέ, στις οποίε επιτρέπεται να συμμετέχουν όλοι οι υποψήφοι και όχι μόνο όσοι έχουν άδεια υποψηφιότητε εκλογέ. Δεν είναι δυνατόν να εκλέγονται όσοι δεν έχουν δημοκρατική εντολή. Επίσης η εντιμότητα, η ελευθερία των εκλογών θα πρέπει να ελέγχεται από ανεξάρτητους παρατηρητές. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους Ιρανούς που είναι φιλιρινικοί και θέλουν ρηξικέλευθες αλλαγές στη χώρα τους. Θέλουν τη διακυβέρνηση από ηγέτες που θα, θα προκύψουν από ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Η κυρία Ρατζαβί ότι αυτό που συνέβη στο Ιράν είναι η αρχή του τέλους του καθεστώτος αυτού. Και έχω κάποιες ελπίδες ότι η κυρία Ρατζαβί έχει δίκιο σε αυτή την πρόβλεψη. Ευχαριστώ. Κύριος Μάριο Μάουρο έχει το λόγο τώρα και σε ετοιμάζεται κύριος Κέλλαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Σουηδική Προεδρία για τις προκαταρτικές, προτακτικά λόγια που είπε. Είπε ισορροπημένα πράγματα για τη συζήτησή μας. Μπορεί να καταλάβουμε ποια είναι η ευθύνη που καλούμεθα να αναλάβουμε. Επιτρέψτε μου εν αυτή τη ενία να κάνω μια παρατήρηση. Αυτή δημιουργείται ε, από αυτά που είδαμε σε όλο τον κόσμο, στις οθόνες των τηλεοράσεων. Δηλαδή τις ε, τα πλήθη που διαμαρτυρόταν. Είναι θεοκρατικό καθεστώς το Ιράν, πράγματι. Και οι ακρεφνείς συνιστώσεις ε, με το πρόσχημα του Θεού εφαρμόζουν τα μέτρα τους. Και είδαμε αυτές τις μέρες τον κόσμο να καταλαβαίνει στις πλατείες και να φωνάζει ο Θεός είναι μεγάλος. Πόση διαφορά όμως. Ε? Στα βλέμματα ε, τη βούληση που εξέφρασαν αυτοί οι άνθρωποι, στην αποφασιστικότητα να μην είναι βίαιοι. Αυτό μας κάνει να καταλάβουμε ότι στο Ιράν η αγάπη για την ελευθερία, για την αλήθεια, η αγάπη για τη μοίρα του λαού, η αγάπη και η προσοχή για τη μοίρα του καθενό δεν είναι κάτι νεκρό. Δεν άρκεσαν 30 χρόνια θεοκρατίας, 30 χρόνια συστηματικής καταστροφής του ανθρώπου για να διαγραφεί αυτή η μνήμη που είναι στην καρδιά όλων μας. Και αυτό θα πρέπει, σε αυτό πρέπει να είμαστε πιστοί. Σε αυτό το γεγονός, την αγάπη για την ελευθερία, την αγάπη για την αλήθεια. Εκεί πρέπει ανεπιφύλακτα να αφοσιωθούμε και θα πρέπει να υπομειστεί ο καθένα τι ευθύνε του. Διότι το να ζητάμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι ισχυρά, να είναι αποφασιστικά, να κάνουν ακουστή η φωνή του, δεν είναι απλή μια γεωπολιτική υπογράμμιση γεγονότων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκπροσωπούν ευρωπαϊκό πρόγραμμα, την Ενωμένη Ευρώπη και θα πρέπει να ανταποκριθούν στην αγάπη ε, για την ελευθερία και την αλήθεια που εκφράζουν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν στους δρόμους τελευταίες ημέρες. Ευχαριστώ κυρία Μάουρα. Και τώρα Κέλλαν, ο επόμενος αγορητής, ο κύριος Κέλλαν, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια σημαντική αλλαγή έλαβε χώρα στο Ιράν. Η πρώτη, το πρώτο μα συμπέρασμα λοιπόν θα πρέπει να είναι ότι το Ιράν δεν είναι και ούτε πρόκειται να είναι ξανά το ίδιο ποτέ γιατί εκατομμύρια Ιρανοί αρνήθηκαν να είναι όμοιροι των ε, ηγετών τους, του κλήρου και απέδειξαν ένα θαυμαστό θάρρος για να αλλάξουν τη δικτατορία. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα δεν είναι οι εκλογές. Αυτή τη φορά προκλήθηκε μια αν θέλετε, διαφυγή για την ε, λαϊκή αγανάκτηση, τόσο μεγάλη που δεν ε, ήταν αναμενόμενη. Και αυτό μου θυμίζει την κατάσταση πριν από 20 χρόνια στην Ανατολική Ευρώπη, όπου κάποιες κυβερνήσεις ήταν ε, προετοιμασμένοι για την πραγματική, για την πραγματική συνύπαρξη με τον κομμουνισμό, αλλά δραστηριοποιήθηκε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και άλλαξε το σύστημα το οποίο και τελικά έπεσε. Γι' αυτό είναι λοιπόν σημαντικό να συνειδητοποιούμε ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση στο Ιράν δεν μπορεί να παραμείνει ίδια. πέρα από τις συνοθείες, τις εκλογές και την καταστολή. Εκτιμάται ότι κατά τα 30 χρόνια δικτατορίας φυλακίστηκαν πάνω από 5 εκατομμύρια άνθρωποι πάνω από 200.000 ε, έχασαν τη ζωή του μέσα από βασανιστήρια και ε, πρόσφατα ότι έχασαν τη ζωή του 200 άτομα τουλάχιστον. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στηρούν πολύ ενδιστακτική στάση και δεν καταδικάζουν αρκετά τα εγκλήματα αυτά. Δεν καλούν το καθεστώς να αναλάβει τις ευθύνες για την συμπεριφορά του. Αν ε, πραγματικά θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των Ιρανών πολιτών, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να βλάψουμε πραγματικά τους δικτάτορες. Και τι εννοώ. Ότι για παράδειγμα θα πρέπει να απαγορεύσουμε την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αποσύρουμε τους διπλωμάτες μας από το Ιράν ως χειρονομία αγανάκτησης. Και να πούμε ότι οι εκλογές μπορούν να λάβουν χώρα στο Ιράν μόνο υπό επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Κολάνσκα Μπομίσκα, κυρία. Κολάνσκα Μπομίσκα έχει το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι. Η κατάσταση χειροτερεύει στο Ιράν. Παραβιάζεται η δημοκρατία. Και αυτό είναι επικίνδυνο για τη σταθερότητα της περιοχής. Πρέπει να εκφράσουμε ανησυχίες και καταδίκη αλλά οι δηλώσει δεν μπορούν να είναι κάτι απλό, συμβολικό και κενό. Κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτε αναφέρονται στην επιβολή νέων κυρώσεων επί του Ιράν. Χρειάζεται όμω συζήτηση τώρα. Τι θα κάνουμε για την πρόθεση της δημοκρατίας σε επίπεδο λαού στην Ευρώπη. Είμαι Πολωνέζα και εμείς στην Ανατολική Ευρώπη ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι δράσεις για την επικράτηση της δημοκρατίας. Έχουμε και εμπειρία στον αφορά την προώθηση της δημοκρατίας στη Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Ευρώπη. Πρέπει να εξετάσουμε τα μαθήματα που πήραμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο Ιράν και τι θα είναι στις παρούσες περιστάσεις αποτελεσματικό για αυτή τη χώρα. Να σας υπενθυμίσω κάτι. Αν θέλει να αξιόπιστη η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να λάβει κάποια μέτρα και στη Μολδαβία σύντομα θα αντιμετωπίσουμε νέο πρόβλημα. Στις 29 Ιουλίου γίνονται εκλογές εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί ούτω ώστε να είναι δίκαιες και ελεύθερες οι εκλογές στη χώρα. Δεν αρκεί να μιλάμε για την υποστήριξη της δημοκρατίας. Εμείς στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είμαστε πιο δραστήριοι σχετικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω κάναμε εξαιρέσεις που δεν μπορούμε να επαναλάβουμε σε αυτό το χρόνο. Δεν μπορεί να παρεμβαίνετε 35 δευτερόλεπτα ε, παραπάνω, όταν σας δείτε χρόνος αγόρευσης ένα λεπτό. Σόνικ, κύριο Σόνικ, ο χρόνος αγόρευσης είναι 60 δευτερόλεπτα, σας υπενθυμίζω. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα, σίγουρα θα πρέπει στο Ιράν να ελεγχθούν ε, οι εκλογές. Αλλά η αρχή της διαθέτησης το, της σύγκρουση αυτής θα πρέπει να είναι μια δήλωση του Ιράν ότι όσοι και απαρνείται τη χρήση βία και καταστολή κατά δημοσιογράφων, διαδηλωτών ή υπηκών ε, άλλων χωρών. Στις, τις οποίες ε, το Ιράν κατηγορεί για την κλιμάκωση αυτής της κατάστασης. Φυσικά θα πρέπει να σεβαστούμε την κυριαρχία του Ιράν, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να θυμίσουμε στις αρχές ε, της Τεχεράνης ότι δεσμεύεται από τις διεθνείς συμβάσεις για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών δικαιωμάτων. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει πυρηνικό πρόγραμμα παρά μόνο για ειρηνικού σκοπού. Θα πρέπει επίση ε, να ανακτήσει την παγκόσμια εμπιστοσύνη το Ιράν και να ε, πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αμυγό ειρηνικό χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κόπα έχει το λόγο. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου λύπη για το τραγικό αεροπορικό ατύχημα που έγινε σήμερα στην επαρχία Κασβίν του Ιράν η σημερινή συζήτηση εδώ είναι επιβεβλημένη μετά τα γεγονότα που ακολούθησαν τις εκλογές της 12ης ιουνίου. θεωρώ όμως ότι πρέπει να τη διεξάγουμε στο σωστό πλαίσιο. δεν πρέπει να δώσουμε λάθος μηνύματα. κάθε άμεση ή έμεση σύνδεση των γεγονότων αυτών με το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος είναι αποπροσανατολιστική. πρέπει να είμαστε σαφείς πως το αντικείμενο της συζήτησής μας σήμερα είναι η κατάσταση της δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο ιράν η φιλολογία επίσης για νέες κυρώσεις δεν βοηθά σε καμιά περίπτωση την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του ιρανικού λαού. η δημοκρατία δεν μπορεί να επιβληθεί με τέτοια μέσα. στην ευρωπαϊκή ένωση οφείλουμε να εντείνουμε τις προσπάθειες για εκδημοκρατισμό και σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών θέτοντας όμως το ζήτημα στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού πολιτικού διαλόγου και δυναμώνοντας τις επαφές μας με την κοινωνία των πολιτών οφείλουμε επίση να ζητήσουμε περαιτέρω διερεύνηση των καταγγελιών για νοθεία στην εκλογική διαδικασία και να τονίσουμε και πάλι ότι το δικαίωμα τη ειρηνική διαμαρτυρία είναι αναφέρετο δικαίωμα των πολιτών κάθε χώρα. πρέπει λοιπόν σήμερα από αυτό το βήμα να καταδικάσουμε περίφραστα τη βία και να ζητήσουμε να εφαρμοστεί έμπρακτα ο σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη έκφραση στο ιράν όπω και σε κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. ευχαριστώ κυρία Κοπά. Ο κύριος Μισελ Γκάλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σωστό, πιστεύω, που κάνουμε στην πρώτη εβδομάδα του καινούργιου κοινοβουλίου τη συζήτηση αυτή. Δυστυχώ, οι πρόεδροι της ομάδα, των ομάδων μα αποφάνθηκαν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρξει ψήφισμα, γιατί ε, εγώ αμφιβάλλω. Νομίζω ότι θα μα βοηθούσε ένα τέτοιο ψήφισμα και θα βοηθούσε και τους αντιφρονούντες στο Ιράν αν είχαμε επιβεβαίωσει τη θέση μας. Αυτά που ως επίσημα δηλαδή ε, αποτέλεσαν το αποτέλεσμα το εκλογικό δεν ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα γιατί οι πιο πολλοί υποψήφοι ε, δεν τους επιτράπηκαν να κατέβουν στις εκλογές δεν είχαν τους ίδιους όρους. Γι' αυτό νομίζω ότι πολιτικά μπορούμε να εξαγάγουμε το συμπέρασμα και να πούμε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αποτυπώνει τη βούληση του λαού του Ιράν. Ας ε, αξιοποιήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα μέσα που έχουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να χρησιμοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών Νομίζω ότι αυτή την πολιτική θα πρέπει βραχυπρόθεσμα να ασκήσουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Ούλριχ Λούνατσεκ. Δεν είναι εδώ. Ε, στην κυρία Ούλριχ. Ευχαριστώ κύριε Προεδρεύοντα, κυρίε και κύριοι. Την προηγούμενη εβδομάδα χάρηκα ιδιαίτερα που ακούσαμε τον κύριο Μαχμαλμπάν έναν Ιρανό σκηνοθέτη, ο οποίος μας είπε με πάσα σαφήνεια ότι πριν από τις εκλογές αυτές το 20% μάλλον η δημοκρατία στο Ιράν ήταν 20% μετά τις εκλογές δεν υπάρχει πλέον καθόλου δημοκρατία στο Ιράν και εγώ ασπάζομαι την άποψη αυτή ήταν πραγματικά μια καταπίεση του δικαιώματο των Ιρανών πολιτών να εκφράσουν τη γνώμη του κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Εμένα με ενδιαφέρει το εξή κυρίω. Στα μέσα Αυγούστου θα υπάρξει μια ε, εκδήλωση για την επανεκλογή σε εισαγωγικά του κυρίου Αχμαντινιτζάντ. Τι θα συζητηθεί στο Συμβούλιο. Θα υπάρξει επίσημη αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκδήλωση αυτή και των κρατών μελών. Ελπίζω να μην υπάρξει επίσημη εκπροσώπηση, γιατί νομίζω ότι μετά από, αυτή την, από αυτές τις εκλογές δεν επιτρέπεται να υπάρξει αντιπροσώπηση των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στάσουμε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου, αλλά νομίζω ότι σε αυτή την εκλογή για το χρήσμα δεν επιτρέπεται να υπάρχει αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ακούσω την ε, δική σας άποψη και τι θα γίνει. Ε, σας ευχαριστώ. Αντώνιο Παντσέρη, επόμενος αγωγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος, όπως ξέρετε, να συζητούμε θέματα εξωτερικής πολιτικής όπως το σημερινό που αφορά το Ιράν με κάποια καθυστέρηση όσον αφορά τα γεγονότα. Όμω, αναφυσβήτητα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν θέλει, μπορεί να δραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την προώθηση της Ευρώπης και του κόσμου να λάβει υπόψη σοβαρά αυτά που συμβαίνουν και να λάβει τις δέουσες πρωτοβουλίες ούτε ώστε του Ιράν να μπορεί να υλοποιηθεί. Πρέπει να αποφύγουμε μετά τη μεγάλη προσοχή που δίνει ο κόσμος μετά τις εκλογές στο Ιράν και τις διαδηλώσεις στους δρόμους που προσπάθησε να καταστήλει βία το καθεστώς στο Ιράν να ακολουθήσει η αποσιώπηση της πραγματικότητας στο Ιράν. Θα πρέπει να δούμε ρεαλιστικό τρόπο τα πράγματα αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφύγουμε το θέμα του Ιράν. Θα πρέπει να δώσουμε τέσσερα προσοχή και εμείς και θα πρέπει και η Σουηδική Προεδρία, που την ευχαριστώ για αυτά που είπε σήμερα, να προωθήσει πρωτοβουλίε ισχυρέ μαζί με τι ΗΠΑ και τη Ρωσία και άλλε χώρε, ώστε να αλλάξει η διαδρομή των πραγμάτων στο Ιράν και ε, θα πρέπει και στα θέματα της δημοκρατίας και επίσης και να έρθει και το θέμα των πυρηνικών. Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη, διότι αυστηρότατα, με κάθε αυστηρότητα τηρήσατε το ένα λεπτό που σας διετέθη. Ο κύριος Βιδαλουγάδρας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τις προηγούμενες εβδομάδες γίναμε μάρτυρες με ιδιαίτερη συγκίνηση της, ε, τα επαναλαμβανόμενα δείγματα ηρωισμού των ε, Ιρανών πολιτών που με γυμνά χέρια προσπάθησαν να αντισταθούν στα ρόπαλα και στα όπλα των ε, θητών τους, των δημίων τους. Κάτι που δείχνει την ε, διακαή επιθυμία των Ιρανών πολιτών για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά η απάντηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ε, μικρόψυχη, άτολμη, αδύναμη. Θα πρέπει να στείλουμε ένα ισχυρότατο πολιτικό μήνυμα προς το Ιράν. Ένα μήνυμα που θα δείχνει την ε, απόλυτη απόρριψη και την καταδίκη για αυτή την θεοκρατική απολυταρχία που επικρατεί στο Ιράν. Και μάλιστα ο Μασού Καρατζάβη, η ηγέτης ε, στο, στην εξορία, το δήλωσε. Θα πρέπει ε, να συγκληθεί μια ανεξάρτητη επιτροπή που θα συγκαλέσει και πάλι ελεύθερες εκλογές υπό διεθνή εποπτεία. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα δημιουργήσει κολυσιεργία και θα παρατείνει αυτή την επονίδιστη κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Κυρία Όμεν Ράιτεν έχει το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω Καλωσορίζοντα τον κύριο Μπίλ, τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ξέρω ότι θα είναι πολύ ε, εντατικοί οι επόμενοι μήνες και θα είναι μεγάλες οι ευθύνε που θα επομιστεί. Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το Ιράν, καταρχάς το καθεστώς είναι πραγματικά κάτι που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, είναι απρόβλεπτο. Κατά δεύτερον, βλέπω ότι έχουν προκληθεί ρήγματα, ρήξεις στο καθεστώς, ιδιαίτερα στο θρησκευτικό μέρος. Κατά τρίτον, διαπιστώνω ότι το καθεστώς, σε ό,τι αφορά τη διαφθορά και σε όλα τα αρνητικά στοιχεία του Πακιστάν και στην Μέση Ανατολή, υποστηρίζονται από το Ιρανικό καθεστώς. Διαπιστώνω λοιπόν ότι ο διάλογος δεν μας βοηθάει, δεν βοηθάει καθόλου. Κατά πέμπτον, διαπιστώνω ότι οι πολίτες, ο λαός θέλουν μεγαλύτερη ελευθερία και δικαίως και θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε εμείς ως Ευρωπαίοι. Πρόεδρε, σας ρωτώ λοιπόν, ρωτώ και εσάς κύριε Προεδρεύοντα, κύριε Μπίλτ, γιατί το Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να προβεί σε πιο σκληρές δηλώσεις και γιατί ακούσαμε μόνο κάποιες χώρες οι οποίες προτιμούν να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους και δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Γκερέιρο Σαλόμ, επόμενος κύριος Γκερέιρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να καταδικάσω φυσικά τα γεγονότα στο Ιράν και την καταστολή και καταπίεση που εφαρμόζει η Ιρανική κυβέρνηση και θα ήθελα να υπερθεματίσω σε σχέση με αυτούς που είπαν ότι θα πρέπει να συνδυάσουμε την πίεση που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διατήρηση του διαλόγου διατήρηση των διαπραγματευτικών διαδικασιών. Γιατί η ιστορία και η πείρα μας έχουν δείξει ότι η ρήξη οποιασδήποτε σχέση, η διακοπή οποιασδήποτε σχέση με αυταρχικά καθεστώτα δεν εξυπηρετεί τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών που υφίστανται αυτά τα καθεστώτα, ενώ ταυτόχρονα αποδυναμώνει τη θέση των προσπιστών της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο πίεσης που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχής γενομένης από τα μέσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέναντι στην Ιρανική κυβέρνηση, στο Ιρανικό καθεστώς, αλλά ταυτόχρονα να κρατήσουμε ανοιχτή τη δίωδο της διαπραγμάτευσης και του διαλόγου, διαλόγου με πιέσεις, μέσω κυρίως του είπα του εκπροσώπου μας Χαβιέρ Σολάνα. Ευχαριστώ. Μάγντι Άλαμ, ο κύριος Μάγντι Άλαμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το Ιράν αντιπροσωπεύει τη βασική απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στον κόσμο, παραβιάζοντας τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και επιδιώκει το στόχο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, απ' την άλλη επαναλαμβάνει τη βούληση να εξολοθρεύσει με φυσικό τρόπο από, να εξαφανίσει το κράτος του Ισραήλ. Η Ευρώπη με τη Σουηδική Προεδρία πιστεύω ότι μπορεί να στείλει ένα σαφές ε, μήνυμα προς το Ιράν. Γενικό μήνυμα λέγοντας ότι οι αδιαπραγμάτευτες ε, αξίες όπως είναι του ανθρώπου, τα δικιά μας τη ζωή, η ελευθερία της επιλογής Όλα αυτά δεν μπορούν να διαχωριστούν από την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων. Και σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο να ξεκαθαριστεί ότι το δικαίωμα για την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ είναι κάτι που δεν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Και η Ευρώπη που γνώρισε το ολοκαύτωμα στο εσωτερικό της δεν θα επιτρέψει να υπάρξει ένα δεύτερο ολοκαύτωμα ε, του κράτους και του λαού του Ισραήλ. Ευχαριστώ. Κύριε Μαγντή Άλαμ, τελευταία παρέμβαση πριν πάρει το λόγο το Συμβούλιο ανήκει στον κύριο Φιλίπ Γιουβίν. Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο για να παρακαλέσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ταχθεί υπέρ της εφαρμογής τεχνικών και οικονομικών κυρώσεων έναντι του Ιράν. Σίγουρα υπάρχουν πολλά επιχειρήματα κατά της επιβολής κυρώσεων, γιατί οι κυρώσεις θα έχουν συνέπειες ε, στη ζωή των Ιρανών πολιτών. Αλλά το χειρότερο για τους Ιρανούς πολίτες δεν είναι η ένδια που θα προκύψει από τις κυρώσεις. Το χειρότερο για τους Ιρανούς πολίτες είναι η σιωπή μας, η αδράνειά μας και η κινησία μας, γιατί οι κυρώσεις δείχνουν το ενδιαφέρον μας και αυτό είναι το σημαντικό. Η Ευρωβουλή πιστεύω ότι οφείλει να απαιτήσει την εφαρμογή κυρώσεων κατά του Ιράν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, ζητήθηκε και άλλη μια παρέμβαση. Μπορώ να τη δεχτώ. Υπάρχει μέγας πλούτος συνεισφορών στο Κοινοβούλιο, κάτι πολύ σημαντικό, διότι είναι πράγματι ευαίσθητο θέμα και ουσιαστικό ο κύριο Τάνοκ για τελευταία παρέμβαση πριν πάρει το λόγο το Συμβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θεοκρατικό, το φρικτό καθεστώς αυτό του Ιράν έχει εγκληματίσει επανειλημμένα. Έχει κρεμάσει ομοφιλόφιλους και 50 αθώους ε, διαδηλωτές τώρα. Δεν θα πρέπει να ε, εκπλησώμεθα διότι ε, διεπράχθη εκλογική απάτη. Πιστεύω ότι έγινε μια ρογμή στο καθεστώς και χαιρετίζω τη διαμαρτυρία των νέων. Νομίζω ότι μπορεί να καταρρεύσει τελικά αυτή η σάπια κυβέρνηση. Ο κ. Χάουιτ σε άλλη συνεδρίαση πρότεινε ότι να, στείλαμε... να στείλουμε παρατηρητέ από το Κοινοβούλιο εκεί για να διαπιστώσουν κατά πόσο πράγματι έγινε νοθείε εκλογέ. Όχι, ποτέ δεν πρέπει να νομιμοποιούμε οποιοδήποτε ψευτοεκλογέ που περιορίζουν του υποψήφιου λόγω θεοκρα... Ε, θρησκευτική αγνότητα και να μετρώνται οι ψήφοι μετά ε, και κλεισμένο των θυρών. Ευχαριστώ κύριε Τάνο και τώρα θα κλείσει τη συζήτηση ο κύριος Μπίλτ, ο εκπρόσωπος ο Προεδρεύων του Συμβουλίου. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο και άκουσα με μεγάλη προσοχή τις διάφορες ε, θέσεις που εκφράσατε και όπως είπατε όντως πρόκειται για μια πολύ σημαντική συζήτηση για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ενωμένοι στην εκτίμησή μας για τα όσα συμβαίνουν, αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις μας και πολύ ε, πιο σημαντικό αυτά που ακούμε από τον κόσμο και επίσης που είναι πιο σημαντικό από αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Θα ήθελα να πω το εξής. Είπατε ότι δεν είμαστε αρκετά σαφείς. Αν θέλετε να κάνουμε συγκρίσεις με τα αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτά που δήλωσαν άλλοι παγκόσμιοι σημαντικοί φορείς, πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εμείς ήμασταν οι πιο συνεπείς, οι πιο σαφείς και οι πιο έντονοι στα λόγια που χρησιμοποίησαμε. Θα θέλαμε τα λόγια αυτά να είχαν μεγαλύτερο αντίκτυπο από αυτό που έχουν. Αλλά αυτό συχνά ισχύει. Ωστόσο, τα λόγια μας δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν σαφή συζητήσαμε αυτά που συνέβησαν στο Ιράν, κυρίως μετά τις εκλογές την 10 η Ιουνίου. Αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε στα όσα είδαμε στις τηλεοράσεις μας και πριν από τον Ιούνιο, γιατί ξαφνικά το Ιράν είχε αλλάξει λίγο από αυτά που είχαμε συνηθίσει. Υπήρχε ένα στοιχείο εντός ε, στα πλαίσια του καθεστώτος πάντα ένα στοιχείο πολυμορφίας, μία επιθυμία για αλλαγή, για μεταρρύθμιση. Αν αυτό αποτύπωνε τώρα την πλειοψηφία των Ιρανών ή όχι, αυτό δεν μπορούμε να το κρίνουμε απ' έξω, αλλά ήταν πραγματικά σημαντική. Σημαντικό το στοιχείο αυτό. Και αυτό διαφαίνεται και από αυτά που συνέβησαν μετά την 12η Ιουνίου. Άρα, καταδικάζοντας αυτά που συνέβησαν μετά τις εκλογές, δεν θα πρέπει να ξεχάναμε το τι συνέβη πριν τις εκλογές και την, ε, αν θέλετε, τον αντίκτυπο των γεγονότων αυτών μακροπρόθεσμα. Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι στις απόψεις μας ο κύριος Αρισβόλψ και ο κύριος Κονπεντήτ, ο κύριος Μάουρα, ουσιαστικά την ίδια θέση υποστήριξαν το πιο δύσκολο όμως φυσικά δεν είναι τα λόγια αλλά οι πράξεις εν ώψη της κατάστασης αυτής και νομίζω θα πρέπει να διακρίνουμε δύο γραμμές. Καταρχάς είναι αρκετά προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι η σαφή φωνή υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις δημοκρατίες παντού, οπουδήποτε και υπό όλες τις συνθήκες. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στην κατάρτιση πολιτικής, αλλά δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρεκκλίνουμε από την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να καταδικάσουμε λοιπόν τις αντικές καταδίκες τους θανάτους. Θα πρέπει να καλέσουμε να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς ε, στην έκκλησή μας για υπέρ της ελευθερίας για κάθε άνθρωπο σε όλο τον κόσμο. Και μπορεί στο τέλος θα πρέπει να υπάρχει ίσως και κάποια διαφωνία, αλλά μπορεί και στο τέλος να χρειαστεί να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε, να λάβουμε δράση. Και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο από το να κάτσουμε και να παρακολουθούμε την κατάσταση. Προφανώς ε, η παρέμβαση είναι κάτι το πιο δύσκολο. Μιλήσατε για τις ιστορικές μας εμπειρίες με τις ε, το γεγονός όμως ότι έχουμε αυτή την ιστορική εμπειρία στην Ευρώπη ίσως και να μας δίνει τη δυνατότητα να αποδηθούμε σε αυτό το δρόμο. Δεν θα πρέπει να πιστεύουμε ότι ο διπλωματικός διάλογος μπορεί να επιλύσει τα πάντα, οποιαδήποτε, όλα τα θέματα τα οποία ακούσαμε σήμερα. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Αλλά δεν ναι, θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία έχουμε καθήκον να εξετάσουμε, να προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε με του διπλωματικού διαλόγου. Και νομίζω ότι οι Γάλλοι φοιτητέ, το διπλωματικό προσωπικό της Βρετανίας υποστηρίζει το διάλογο. Προέρχομαι από μια χώρα που το 1% του πληθυσμού έχει εμπειρία από το Ιράν και μετακινείται συχνά στο Ιράν. Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να παρέμβουμε για να βοηθήσουμε συγκεκριμένα άτομα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρίς να πιστεύουμε ότι αυτό πρόκειται να επιλύσει, να επιλύσει όλα τα ζητήματα. Και έχουμε και το πυρηνικό θέμα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι υπάρχουν απλές λύσεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιαδήποτε λύση αν δεν ξεκινήσουμε πραγματικό διπλωματικό διάλογο. Και θα πρέπει να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Και προφανώς αυτό θα καταστεί ακόμα πιο δύσκολο στις σημερινές καταστάσεις. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπό αμφιβολία. Και ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα κάποιες από τις δύσκολες επιλογές και κάποιες από τις δύσκολες κρίσεις τις οποίες θα πρέπει να προβούμε τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Όχι όμως παραπάνω από αυτό. Και όλοι θα πρέπει και εσείς και εμείς στο Συμβούλιο να δραστηριοποιηθούμε μαζί με άλλους παγκόσμιους φορείς και με την ε, κυβέρνηση Ομπάμα αλλά και με άλλους, με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τη Ρωσία, με την Κίνα και με την ευρύτερη ε, παγκόσμια κοινότητα γιατί μόνο από κοινού μπορούμε να ξεκινήσουμε την επίλυση όχι μόνο των κατεπηγόντων θεμάτων αλλά και άλλων θεμάτων τα οποία θα πρέπει να επιληθούν. Σας ε, είμαι ευγνώμων λοιπόν για τη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι υπογραμμίστηκε η σαφή ομοφωνία που επικρατεί σε ό,τι αφορά την προάσπιση των αξιών μας, αλλά και ότι τονίστηκαν κάποιες από τις δύσκολες επιλογές, ε, τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε τους επόμενους μήνες. Ξέρουμε τι θέλουμε να πετύχουμε και ότι θα πρέπει να το επιδιώξουμε. Αλλά μην φανταστείτε ότι θα είναι κάτι το εύκολο και θα σας διαβεβαιώ, σας ότι το Συμβούλιο θα συνεχίσει να ασχολείται με όλες τις πτυχές του θέματος αυτού. Ευχαριστώ πολύ το Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν είναι σημαδιακό ή όχι ότι οι πρώτες μου λέξεις... Ναι, κύριε Κομπέντετ. Συγγνώμη, αλλά μόλις έλαβα μια πληροφορία και θα ήθελα να τη διαβάσω στο Συμβούλιο και στους συναδέλφους. Η Νατάλια Στιμήραβα, που ήταν ε, υποψήφια για το βραβείο Ζαχάροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνελήφθη το πρωί στον Κρόσνη. Απήχθη στον Κρόσνη από άγνωστους απαγωγείς και θα ήθελα να ζητήσω από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για να μάθουν στη Μόσχα ότι σκεφτόμαστε την Νατάλια Σεμίροβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κομπέντη. Είμαι βέβαιος ότι το Συμβούλιο όπως και ε, το Κοινοβούλιο ε, λαμβάνει υπόψη αυτό που είπατε και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Η συζήτηση έληξε η προηγούμενη και έχει ζητήσει επί προσωπικού ζητήματος αν με το λόγο ο κύριος Χάουιτ. Ε, το παρέθεσα το όνομά μου ο κύριος Τάνοκ, ότι είπα κάτι. Στη συζήτηση ήμουν σαφέστατος. Είπα ότι αν οι περιστάσεις το δικαιολογούσαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν σε θέση να στείλει παρατηρητές στις εκλογές του Ιράν. Αλλά ακριβώς επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πίστευε ότι μπορεί να το κάνει, ε, Μπορούμε να αμφισβητούμε τη εξαγωγή αυτών των εκλογών. Λυπούμε ότι ο κ. Στάνοκ δεν τα άκουσε σωστά όταν τα ανέφερα. Ήθελα απλώ να διορθώσω αυτή την εντύπωση που σχηματίστηκε. Ευχαριστώ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την Κίνα. Ε, τον ε, λόγο εξ του Συμβουλίου ε, έχει ο κύριος Κάρλ Μπίλτ. Κύριε Μπίλτ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, άλλη μια συζήτηση